Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να σας ε, ρωτήσω. Η έρευνα του Κοινοβουλίου για την απάτη ε, με την ψηφοφορία ε, που έκανε διέπραξε η κυρία Λεπέν. Πώς προχωρά αυτή η έρευνα. το σώμα θα ενημερωνόταν για το αποτέλεσμα, για το αποτέλεσμα είχαμε πληροφορηθεί. Θα ήθελα Επίσης να σας πω ότι ένα μέρος αλήθειας ε, έχει ε, συγκαλυφθεί διότι ο συμπρόεδρος Μαρσέλ Ντεγκράφ ε, λέει η κυρία Λεπέν ψήφισε στη θέση της αλλά παρέλειψε και έκρυψε από εμάς ότι και ο Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Μετόπου ο κύριος Νικολά Μπέι επίσης ψήφισε για λογαριασμό της κυρίας Λεπέν και συγκεκριμένα την ομοθεσία για την υπόθεση Volkswagen και τις εκπομπές αερίων. Σας παρακαλώ να λάβετε υπόψη στην έρευνα του Κοινοβουλίου και αυτή τη δεύτερη απάτη, άρα και από τον Συμπρόεδρο και από τον Γενικό Γραμματέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Σας ενημερώνω ότι ο πρόεδρος που διερευνά το θέμα και ένα διαδικαστικό τώρα, η κυρία Λεπέν. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία για να δοξαστεί η συνάδελφος. Αλλά βάσει το άρθρου 22, εδάφιο 4, και δυστυχώς θα αναγκαστώ να ε, αντιστρέψω τους δαυλούς και τους χρυσούς της δόξα σας ε, και να σας δείξω ε, την πραγματική οδό γιατί ξεχνάτε την πραγματικότητα της εγχειρίας του περασμένου πολέμου, το τέλος του πολέμου που οδήγησε σε 9 εκατομμύρια θανάτους στην Ευρώπη για τον Πρώτο Παγκοσμίο Πόλεμο θα έπρεπε να σέβονται οι ευρωπαϊκοί θεσμοί την αργία των ημερών που ε, τους φιλοξενούν. Γαλλία και Βέλγιο. Θα έπρεπε να ε, γίνεται ε, και να σεβαστώ αυτό το καθήκον μνήμης και ως δείγμα διαμαρτυρίας ζητώ από τους Γάλλους να εγκαταλείψουν το επικύκλο και να μην συμμετάσχουν στις ψηφοφορίες. Διαδικαστικό. Κύριε Πρόεδρε, τουλάχιστον δεν θα έχουμε για μια φορά απάτη με την ψηφοφορία, αφού θα φύγουν όλοι από την αίθουσα. Καλό αυτό επομένω. Μπορούμε τι θα γίνει με την περίπτωση νοθείας. αλλά και τι θα κάνουμε με τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών εδώ, εάν υπάρξουν ε, ψηφοφορίες που το αποτέλεσμα θα κρυθεί για μία ψήφο διαφορά, λόγου χάρη. Θα το δούμε. Ε, διαδικαστικό και πάλι. Κύριε Μπερμάγερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν έγινε κάποιο μεταφραστικό λάθος. Ίσως εγώ δεν άκουσα καλά, αλλά κάποιο εξέφρασε την ικανοποίησή του που κάποιο άλλο αντιπαθητικό έφυγε από το ημικύκλιο. Νομίζω όμω ότι εδώ οφείλεται συγγνώμη και είναι ντροπή ε, εσεί, ε, ο πρόεδρο, να παίρνετε μια τέτοια θέση. Ιδάλω υπήρξε μεταφραστικό σφάλμα. Όμω, αν είπατε αυτό που μου φάνηκε, οφείλεται συγγνώμη. I think the wrong translation. Νομίζω ότι έγινε λάθος στη μετάφραση. Διαδικαστικό. Ο κύριος Μελανσόν. Κύριε Πρόεδρε, είμαι Γάλλος. Δεν θα φύγω από το Εμικύκλιο γιατί σέβομαι το σώμα της Ολομέλειας. Όμως να ξέρετε ότι η μέρα αυτή ξεκίνησε με χιλιάδες ε, εορτασμούς της επαιτίου από την το τέλος ε, των ε, επανελειμμένων σφαγών που οργανώθηκαν σε αυτή την Ήπειρο κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Ελπίζω να μην ξαναδούμε ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο τα όσα προηγήθηκαν στις 11 Νοεμβρίου. Και ελπίζω αυτό να το θυμάμαστε όλοι και να το σεβόμαστε. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε όμως τώρα στις ψηφοφορίες. Έχουμε την έκθεση Ζωρίνιο για τις λύσεις διαλειτουργικότητας ως μέσο εξυγχρονισμού του δημόσιου τομέα. Από την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Περνάμε στην ψηφοφορία. Okay. 1. Ε, Ψηφίζουμε συνολικά το κείμενο, μπλοκ 1, τροπολογία 92, ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ονομαστικά τώρα το ψηφίζουμε την πρόταση Κομισιόν της ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στην ψηφοφορία. Επί του νομοθετικού ψηφισματός με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και το ψήφισμα θετικού περιεχομένου. Σας ευχαριστώ. Και τώρα πρενούμε στην ε, ψηφοφορία της Μελλοντικής δέσμης για τις αεροπορικές μεταφορές σχέδιο σε σε 1, αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 3 αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 4, αρχικό κείμενο, πρώτο τμήμα ψήφι ΠΕΡ, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ψήφι ΠΕΡ, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 5, αρχικό κείμενο, ψήφι ΠΕΡ κατά αποχές εγκρίνεται σε 6 αρχικό κείμενο ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Παράγραφο 7 αρχικό κείμενο δύο τμήματα πρώτο ψήφι πέρ κατά αποχές εγκρίνεται Δεύτερο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 8. Αρχικό κείμενο. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 11. Αρχικό κείμενο. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 12. Αρχικό κείμενο. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ψήφι ΠΕΡ. κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 15 αρχικό κείμενο ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 16 αρχικό κείμενο ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 17, αρχικό κείμενο, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και με μεγάλη πλειοψηφία. Μετά την παράγραφο 17 έχουμε μια προφορική τροπολογία. Ο συνάδελφος ε, κ. Μαλτέζ. Το κείμενο καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την προστασία των εργαζομένων και των καταναλωτών σε περίπτωση πτώχευσης μιας εταιρείας μεταφορών. Εδώ χρειαζόμαστε εξηγήσει σε σχέση με ήδη με περιστατικά που έχουν ήδη συμβεί και με μελλοντικέ περιπτώσει. Ευχαριστούμε. Πέρα αυτή τη τροπολογίας. Έχουμε μια νέα κατάσταση εδώ. Πρέπει να μετρήσουμε τους συναδέλφους που σηκώνονται για να στηρίξουν την τροπολογία και αν είναι 40 ή όχι. Είναι δεν είναι 40 δυστυχώ συνάδελφοι, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε για την και τροπολογία λοιπόν. Γι' αυτό θα ψηφίσουμε το αρχικό κείμενο. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 19. Αρχικό κείμενο. Ψήφι υπέρ. Να σηκώνετε καλά τα χέρια. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 20. Αρχικό κείμενο. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 21. Αρχικό κείμενο. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 22 αρχικό κείμενο κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 23 αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ. αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 26 αρχικό κείμενο δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται παράγραφος 27 αρχικό κείμενο δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 28 αρχικό κείμενο ψήφι υπέρ αποχές εγκρίνεται. Θεολογική σκέψη F κείμενο ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πολύ καλά, θέλετε να ελέγξουμε, άκουσα. Να ελέγξουμε, άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ε, Προχωρούμε λοιπόν. στην ψηφοφορία της εκθέσεως ε, Χούμπνερ και Λάινεν για τη μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Ψηφίζουμε αρχικά μια δέσμη τροπολογιών. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 12. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Ονομαστική και αυτή η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 26. Τροπολογία 50 από το νόμο το πράσινο, επίσης ονομαστικά έρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 63 από ΕΛΚ, Σοσιαλιστές Δημοκράτες και ΑΛΔΕ, ονομαστικά άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 35 από το Μαδάλντε. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστικά, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. zamknięte. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 51 καταπίπτει και περνάμε στην τροπολογία 3. Ψηφίζουμε ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 42. Καταπίπτει. Περνάμε στην τροπολογία 7. Ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Πάντως πρέπει να πάμε λίγο πιο πίσω. Στην τροπολογία 42 που με ενημερώνουν πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία. Δύο τμήματα εδώ, τροπολογία του ΕΛΚ, η 42 λοιπόν. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πού πάμε. Τροπολογία 43 του ΕΛΚ σε τρία τμήματα. Ονομαστικά το πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα επίσης ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Το τρίτο τμήμα ονομαστικά ψηφίζουμε άρχεται η ψηφοφορία. θέλει κάτι να πει. Uh, uh, Πρόεδρε, δεν έχει κανένα νόημα αυτό το τρίτο κομμάτι. Στο το 2024 δεν θέλουμε να έχουμε ισότητα των φίλων. Αλλά νωρίτερα. Αυτό θέλαμε να ψηφιστεί για νωρίτερα. Γι' αυτό το καταψηφίζουμε το 2024. is correct, has been right. Καλά τα είπατε. Τροπολογία 6 τώρα. Καταπίπτει πηγαίνω στην τροπολογία 52 πράσινη ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Α, μου λένε όμως ότι καταπίπτει και 52, άρα ψηφίζουμε την τροπολογία, υπάρχει μόνο 8, ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 8. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Ψήφι περ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 53. Καταπίπτει. 54. Επίσης. τροπολογή 22 τώρα. Ψηφίζουμε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 55. Και περνάμε στην 41. Έλξος Ιστές Δημοκράτης. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. 56 και 57. Α, καταπίπτουν. 58 επίσης καταπίπτει. Ψηφίζουμε την 28. Ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφο σε ένα αρχικό κείμενο. Πέντε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται τρίτο τμήμα ονομαστικά άρχεται ψηφοφορία Πέραση zostaje Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα, ψήφι περ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πέμπτο τμήμα, ψήφι περ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2, τροπολογία 61, ECR, ψήφι περ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο παραγράφου 2, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 4, αρχικό κείμενο, ονομαστικά, άρχεται ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 5 αρχικό κείμενο, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ονομαστικά. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστικά. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 6. Αρχικό κείμενο κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται μετά την παράγραφο 6 τροπολογία 45 α, πίπτη, παράγραφος 7 64 D τροπολογία ονομαστικά ψηφίζουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται Παράγραφος 8, αρχικό κείμενο. Ονομαστική ψηφοφορία, Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 9. Καταπίπτει τροπο 46, οπότε ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο της 9 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα ονομαστικά τώρα. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα. Μετά την παράγραφο 9, τροπολογία 47 των πρασίνων ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ε, Καταπίπτει η επόμενη 44D. ΕΛΚ. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 17, αρχικό κείμενο. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 20, αρχικό κείμενο, σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία ονομαστική. Υπέρ. Συγγνώμη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 49. Γιατί καταπίπτει 22 των πρασίνων. Περνάμε στην 22 αρχικό τμήμα. Πρώτο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Και εδώ ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 24 αρχικό κείμενο. Ονομαστική ψηφοφορία έρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Αιτιολογική αναφορά 4, αρχικό κείμενο, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Μετά την αιτιολογική και αναφορά 7, 62, ΕΛΚ και Δημοκράτες. Υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνατε. Είναι αργά, έχει περάσει η ώρα, αλλά σας παρακαλώ να σηκώνετε ψηλά τα χέρια σας για να το βλέπουμε. Αιτιολογική σκέψη Α, σε δύο τμήματα, από το τμήμα, υπέρ. Θα πάτε καλύτερα τώρα. Κατά. Αποχές. Εγκρίνατε. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη Β. Αρχικό κείμενο, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Αιτιολογική σκέψη Ε. Τροπολογία 36. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Ιδεολογική σκέψη F, σιγματάφ. Υπέρ, κατά. ποιες εγκρίνεται. 33 των ζωτερικών και μεταρρυθμιστών, ονομαστική. Υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Τη σκέψη J. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. L37. Για τα β δηλαδή. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ε, ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Και πάλι L, δεύτερο τμήμα για το αρχικό κείμενο. Ε, υπέρ, κατά. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη M59 των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο, πάλι εμ, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Νη, αρχικό κείμενο, πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Ναι. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται νομίζω. Αιτιολογική σκέψη ο αρχικό κείμενο, ε, ονομαστική ψηφοφορία άρχεται, για τα ε δηλαδή, πέρας. Ανεβαίνει η αγωνία για περιμένω το αποτέλεσμα, εγκρίνεται. Τώρα, 34 ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας. Εγκρίνεται. Q32. Q δηλαδή για τα ζήτα. Ε, των συντεχνών των άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Αρνητικό αποτέλεσμα. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη Q. Αρχικό κείμενο. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Προσοχή. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Περιμένουμε το αποτέλεσμα. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη έ ε, Ι. Ήτα τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη τι τάπα σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ε, υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία μάλλον ονομαστική πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα και εδώ ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας, εγκρίνεται. Γιου, 60 των συντηρητικών και αριθμιστών, 60 δηλαδή ΚΑΠΑ. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 38 της ΕΝΕΦ. Ονομαστική ψηφοφορία έρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Γιούσε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα τώρα, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη ΚΒ. 39. ενεφ, Άρχεται η ψηφοφορία, ονομαστική. Πέρας. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορια τερας Πέρας. Εγκρίνεται. W40, τα παγάμα δηλαδή, ENF, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. W και πάλι καπαγάμα, αρχικό κείμενο, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. X, κάπα αρχικό κείμενο, ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη ΑΑ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Αποτέλεσμα εγκρίνεται. Επί τέσσερα τμήματα. Ε, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τέταρτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αιτιολογική σκέψη ΑΑC ΚΑΠΑ θ ονομαστική ψηφοφορία άρχεται ε, πέρας Πρόλαβα, λέει ο πρόεδρο. Εγκρίνεται. AD, αρχικό κείμενο. Λάμδα δηλαδή υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. AF, λάμδα β δηλαδή αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη. AG, λάμδα γάμα αρχικό κείμενο. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά. Ας επαληθεύσουμε εδώ. Διότι εδώ δεν είναι σαφής, σαφές το αποτέλεσμα. Ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα. Περνάμε στο AH, λάμδα δέλτα, αρχικό κείμενο, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου, το σύνολο του κειμένου ψηφίσματος που τροποποιήθηκε, ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ όλους και όλες. Καλή σας όρεξη για όσους μπορούν να να φύγουν για το δείπνο. Σας ζηλεύω λίγο, μάλλον σας ζηλεύω πολύ. Thank you, President. Very good. <laughs> Um, we, have a little pause now. Yeah.